Okay. λοιπόν στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Χαίρομαι που βλέπω και νέα μέλη που δεν έρχονται ποτέ στην Επιτροπή. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη γι' αυτό. Παρακαλώ καθίστε αμέσω και ησύχω για να ξεκινήσουμε. Και να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη γρήγορα και αποτελεσματικά. Έχουμε ήδη κάποιους εκ των αναφερόντων. Λυπάμαι που θα πρέπει να περιμένετε λίγο, γιατί πρέπει να γίνει και μια ψηφοφορία και να τελειώσουμε με τα τυπικά και μετά θα έρθει και η σειρά σας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη συνεδρία της Επιτροπής Αναφορών και ελπίζουμε να έχουμε ε, μια γόνιμη πρωινή συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν ε, ενστάσεις, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και σημειώνουμε και ότι η απογευματινή συνεδρίαση σήμερα θα ξεκινήσει στις 2.30. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν 2.30 το απόγευμα. Είναι μια συμφωνία για μια δοκιμαστική ε, προσπάθεια για όλες τις επιτροπές. Έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ περιορισμένες οι διάφορες ε, χρονικές προθεσμίες και για να μπορούμε να διεκπαιρεώνουμε τα θέματα έχουμε μισή ώρα επιπλέον. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι και πολύ θετικό. Να φάτε στα γρήγορα λοιπόν και να επιστρέψετε στις 2.30. Πάμε στο σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Ιουλίου, 10 και 11 Ιουλίου. Σας έχουν διανεμηθεί και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Ωραία. Και θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι θα θέλαμε να καλωσορίσουμε μια νέα ε, ασκούμενη στην γραμματεία της ΠΕΤΗ, η Τεοχάνα Εγνάτοβα. Πού είστε? Ωραία, καλωσορίσατε είναι από τη Βουλγαρία και θα εργάζεται μαζί μας εδώ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Προσβλέπουμε λοιπόν στη συνεισφορά σας και θέλω και να μερίσετε και πώς σας καλωσορίσανε και αν έχετε και δουλειά και ουσιαστικά πράγματα να κάνετε. Ε, είμαι βέβαιη ότι θα βοηθήσετε ιδιαίτερα και τη γραμματεία και εμάς. Δεν έχουμε τίποτα υπό τα διάφορα, δεν έχει θέσει κανείς κάτι, επομένως μπορούμε να περάσουμε απευθείας στην ψηφοφορία για την ετήσια έκθεση για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Έκθεση για το 2016. Η συγκήτρια είναι η Μαρλέν Μίτσι, είναι εδώ μαζί μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε δύο λόγια πριν ψηφίσουμε. Όχι, ευχαριστώ. Ήταν πολύ καρποφόρες οι συνεδριάσεις με τους κοιόδης Θεωρώ ότι η έκθεση είναι καλή. Ελπίζω λοιπόν να πάνε όλα καλά και ευχαριστώ τους και οδησιητές και τους βοηθούς. Okay, I hope that you have your voting cards. Ελπίζω να έχετε και τις κάρτες σας στα μηχανήματα. Όχι, καλό είναι και η συγγήτρια να βάλει την κάρτα της ε, στο μηχάνημα. Και τώρα... I'm not waiting for anybody. Δεν περιμένω κανέναν. Ξεκινάει η ψηφοφορία αν δεν είστε εδώ εγκαίρως, πρέπει να υποστείτε και τις συνέπειες. Λοιπόν, παράγραφος 3. Υπέρ. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασ... Τροπολογία 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική να κάνουμε μια επαλήθευση για την 37. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 37. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται συμβασική τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 48 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 αποσύρθηκε. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 Υπάρχουν ενστάσεις στην προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Κατά της προφορικής τροπολογίας πρέπει να το επαληθεύσουμε. First, vote for the first part in favor. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία, η ηλεκτρονική επαλήθευση της 73. And the vote is now closed. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 κατά τμήματα ψηφοφορία το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα το σύνολο της έκθεσης. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με ευρία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Συγχαρητήρια επίσης ε, στην Ευρωπαϊκή Διαμεσολαβήτρια που κάνει εξαιρετική δουλειά και με αυτήν την έκθεση ε, θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η εργασία της. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, ώστε όσοι πρέπει να αποχωρήσουν την αίθουσα να το κάνουν αυτό ε, πολύ γρήγορα και ήσυχα. Fine. So, λοιπόν, λοιπόν, όλοι οι παρασημοφορημένοι φιλοξενούμενοι μας παρακαλώ να καθίσουν για να ξεκινήσουμε. 1468 περιβαλλοντικές επιπτώσεις ε, για την ε, οικοδόμηση ενός αυτοκινητοδρόμου σε σεισμογενή περιοχή και η 18 του 17 Μιραντολέζη, χώρος Natura 2000 και άλλη μια περιοχή στην Εμίλια Ρωμάνια που φύγεται επίσης από τον αυτοκινητόδρομο. Καλωσορίζω λοιπόν και τους δύο και δίνω το λόγο στον Λούκα Φεριόλη. Για λίγα λεπτά, τρία λεπτά, τέσσερα παρακαλώ. και μετά ο Σιλβάνο τα λιαβάνει μάλλον. Πρώτα όμως θα πάρει το λόγο ο κ. Σφαιριόλη. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν έχω πολλά λεφτά στη διάθεσή μου, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να υπογραμμίσω τα κρίσιμα σημεία της υπόθεσής μας. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Οι οδικές υποδομές είναι σημαντικές για μια περιοχή σαν τη δική μου και έχει μεγάλη σημασία η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία φυσικά των ανθρώπων που ζουν εκεί. Μια επιπόλαια δραστηριότητα στον τομέα των δημοσίων έργων προκαλούν προβλήματα ε, κυρίως στην οικονομία. Αλλά αυτά αποκαθίστανται, αλλά οι βλάβες στο περιβάλλον και οι βλάβες στην υγεία είναι δύσκολο να αναστραφούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει και στην απόφαση ε, που οδήγησε στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την ε, βιοπικιλότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές βλάβες. Αυτό θα πρέπει να βοηθήσει να πετύχουμε τον βασικό μας στόχο της 26ης Μαρτίου του 10 να σταματήσουμε την απώλεια της βιοπικιλότητας μέχρι το 2020. Επίσης υπάρχει και το άρθρο 35 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την Προστασία της Υγείας. Λέγεται ότι πρέπει να υπάρξει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και το άρθρο 37 λέει ότι το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι συμβατή με την αρχή της αηφόρου ανάπτυξης. Έχουμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα κατασκευής αυτοκινήτων δρόμων ασύμβατο με την κατάσταση η οποία επικρατεί. Φύγονται γεωργικές περιοχές υψηλής ποιότητας, υπάρχουν συνέπειες στο κλίμα, υπάρχει ηχητική μόλυνση, παραβιάζονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση με το θόρυβο και αύξηση των κινδύνων για τους υδάτινους πόρους και την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε σύμφωνα με το 2143 και 2017-030 με συνέπειες για τα επίπεδα υγείας και ζωής των πολιτών όπως ακριβώς ε, περιγράφονται στην ανακοίνωση τύπου της 27ης Απριλίου του 2017. della direttiva sugli appalti in house, considerando che ad oggi la società Autobrenner SPA και Υπάρχει ένα θέμα επίση και με τον τρόπο με τον οποίο ε, δίδονται, ε, παραχωρούνται οι άδειε για την κατασκευή των έργων αυτών των οδικών. Είναι ασύμβατε οι μέθοδοι που ακολουθούνται από την επιχείρηση Autobrenner Spa η οποία έχει το 51% του συνόλου των εργολάβων που είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή και η κατασκευή ως προβλέπεται τώρα θα οδηγήσει σε νέα πρόστιμα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βλάβες μπορεί να είναι ε, πραγματικά ανεπίστρεπτες και να δημιουργήσουν ένα παράδεκτο προηγούμενο που δείχνει ότι πληρώνοντας ένα μικρό πρόστιμο μπορεί κανείς να παραβιάζει όλους τους κανόνες. Η οδηγία αυτή λοιπόν δεν γίνεται σεβαστή σε εθνικό επίπεδο στη συγκεκριμένη περίπτωση και θα μπορούσαν να υπάρξουν άλλες λύσεις με την ενίσχυση του σιδεοδρομικού δικτύου το οποίο ήδη υπάρχει και το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί ή την ε, διεύρυνση της εθνικής οδού. Ευχαριστώ, τελειώσατε με κομψό τρόπο και θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ταλιαβιάννη, να πάρει το λόγο και αυτός μέχρι πέντε λεπτά, όχι περισσότερο. Δεν είχατε τελειώσει, συγγνώμη, νόμιζα ότι τελειώσατε διότι ούτως ή άλλως έχετε περάσει τα 5 λεπτά σα. Θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε σε 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Θα διαβάσω λοιπόν τις τελευταίες γραμμές του μηνύματος μου. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ναι μεν αυτός που μολύνει πληρώνει αλλά όχι ότι αυτός που πληρώνει έχει δικαίωμα και να μολύνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το λανθασμένο μήνυμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει χειροτέρευση των συνθήκων υγείας, υπάρχει αύξηση της θνησιμότητας και 83 παραβάσεις υπάρχουν από πλευράς των επιχειρήσεων αυτών, οι 18 αφορούν το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ που επισημάνατε σαφέστατο ότι έχουμε την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει που θα πρέπει να εφαρμόζεται. Εξαιρετικά. Τώρα να δώσω το λόγο στο συνάδελφό σας το πολύ 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, η έκθεση αυτή έχει στόχο να δείξει λίγο ευρύτερα τα όσα κατήγγειλε και ε, η ε, αναφορά και πιο συγκεκριμένα ε, περιβαλλοντικές συνέπειες αυτής της κατασκευής η οποία εάν υλοποιηθεί θα έχει συνέπειες σε όλο το τοπικό οικοσύστημα σε πολύ μεγάλη περιοχή λόγω και της γεωγραφικής του έκτασης. Δείτε το παράρτημα 1. Το σχέδιο του αυτοκινητοδρόμου Τσις Παντάνε, που είναι κατηγορία Α, έχει πολύ σοβαρές ε, συνέπειες ε, για έναν ε, ταχύ αυτοκινητόδρομο κατηγορίας 5. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο αυτοκινητόδρομος που έχει χαραχθεί αφορά την αστική περιοχή. Και ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό είναι γιατί ε, βρίσκεται σε κατοικημένες περιοχές. Το σχέδιο είχε ήδη φτάσει σε τελική λύση το 2004 και αυτό θα είχε λύσει με πολύ μεγάλες και αποταμιεύσεις ε, πολύ σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας ε, κυρίως όσον αφορά το τοπικό παραγωγικό σύστημα, το οποίο είχε πολύ μεγάλη ανάπτυξη μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά και πρέπει να υπάρχει σύνδεση ε, μεταφοράς εμπορευμάτων και ατόμων και να λάβει υπόψη τους και την παραγωγική δομή των ενδιαφερομένων. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία παράγονται εκεί, όπως για παράδειγμα το παρεμετζάνο-ρετζάνο και άλλα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, βιολογικών και, προ... και pop. Όσον αφορά τώρα τη σύνδεση με το παγκοσμιοποιημένο σύστημα μεταφορά ατόμων και εμπορευμάτων ε, μέσω και ε, μεγάλων αποστάσεων, θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικέ ε, μεταφορές ε, μέσω σιδηροδρόμων ή μέσω ναυτιλίας όπως ζητάμε από το 2002 και το είπε και τα επόμενα χρόνια η Επιτροπή Μεταφορών στην τετραετή της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραρτήματα 1 και 2 οι υποδομές ε, των αυτοκινητοδρομών ε, της Παντάνε περιλαμβάνεται σε ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο το οποίο είναι ήδη πάρα πολύ επιβερημένο, παράρτημα 3α και 3β και κυρίως τα αίτια είναι η γεωγραφική θέση διότι βρίσκεται στο επίκεντρο της κοιλάδας της Παδανίας και για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, κυρίως το χειμώνα, υπάρχει πλήρης απουσία ε, ρευμάτων και έτσι διακόπτεται η κυκλοφορία του αέρα και ρηπαίνεται η περιοχή υπάρχει και σχετικό παράρτημα. Είναι ε, βιοτέχνες και γεωργοί κατά βάση οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά δεν υπάρχει καμία συνέχεια από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά ε, και ε, ακριβώς για αυτό το πλαίσιο, βλέπετε και παράρτημα 5, στα σύντο χρόνο δημιουργήθηκε μια κατάσταση ε, στο αέρα, η οποία είναι καταγεγραμμένη με σε πολύ σημαντικό βαθμό και υπάρχουν και καταγγελίες στον τύπο υπάρχουν δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράρτημα 6 και άλλες πηγές, παράρτημα 7. Με την υλοποίηση αυτής λοιπόν της ε, ε, νέας ε, αρτηρίας θα υπάρξουν αρκετά φορα... περισσότερα προβλήματα, θα περνούν βαρέα οχήματα και η κίνηση φυσικά θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο και θα υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Ε, υπάρχει και σχετική περιβαλλοντική εκτίμηση επιπτώσεων και ε, υπάρχουν θέματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα και έχουν καταγγελθεί επανειλημμένως. Υπάρχει ανάγκη να αντιστραφούν οι τάψεις αν θέλουμε να σεβαστούμε και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ποιότητα του αέρα για πιο καθαρό αέρα στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο θέμα υγείας ανθρώπων εδώ. Ήδη από τώρα όλο το οικοσύστημα σε ένα ευάλωτο περιβάλλον ε, έχει πρόβλημα και μόνο χάρη στο Natura 2000 καταφέραμε να διασώσουμε αυτό το οποίο είχε παραμείνει. Ε, υπάρχει ένα σύνολο καναλιών και παραποτάμων και τον οπάδος ποταμός ε, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες ε, πλήττονται εδώ και αυτό το σύστημα θα επιβενεθεί πολύ περισσότερο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και όταν θα κατασκευαστεί ο νέος αυτοκινητόδρομος ε, της Παντάνα. Και υπάρχουν ε, και μικρά τοπικά προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το ε, οικολογικό περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο τα οποία θα επιβαρυνθούν πάρα πολύ. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο αντιτίθεται στους βασικούς στόχους που έχει η ίδια η περιοχή της Εμίλια Ρουμάνια. Και ε, υπάρχουν αποδείξεις για τα όσα σας είπα, υπάρχουν περιγραφές που αποτελούν ε, τμήμα της ε, ε, θετικής έγκρισης που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θάλασσας και υπάρχουν 57 γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Επαλήθευσης του Περιβάλλον, 127 από την περιοχή της Εμίλια Ρωμάλια και 8 από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε πολλές περιγραφές που περιλαμβάνονται ζητήθηκε από την περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια και ε, να λάβει τα μέτρα της και θα ήθελα να ζητήσω και μερικά ε, δευτερόλεπτα για να εκφράσω και μία απορία, μία δυσκολία σε μέσω κάποιων ερωτήσεων. Πώς είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο θέμα ε, με συγκεκριμένη βιοποκυλότητα στην περιοχή η οποία βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε ιστορικό επίπεδο, λόγω των συνεπειών και υπάρχει σύνδεση μόνο μέσω πολύ μικρών διαδρόμων και σε όλη τη διαδικασία της ανάλυσης δεν ελήφθη υπόψη η μελέτη η οποία θα έπρεπε να είχε γίνει ευθύ εξ αρχής ε, στο συγκεκριμένο ε, έργο ε, και έγινε μόνο στο τελικό επίπεδο και όχι σε προκαταρκτικό στάδιο. Πώς είναι δυνατόν η Επιτροπή Βία να αποφάσισε να δώσει τη συγκατάθεσή της για την κατασκευή αυτού του αυτοκινητοδρόμου όταν υπάρχουν όλα αυτά. Και με αυτά τελείωσα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία και να τα ζητάμε από δήμους που δεν έχουν ανθρωπίνους, τεχνικούς αλλά κυρίως οικονομικούς ε, πόρους για να κάνουν αυτές τις αναλύσεις. Ζητώ από την Επιτροπή σας να αφήσει ανοιχτή αυτή την αναφορά για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητο, να εμβαθύνουμε και να μπορέσουμε να λάβουμε ε, την κατάλληλη απάντηση από εσά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, προσοχή σας και σας εύχομαι και καλή δουλειά. I Σας ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Τσιπριάνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξετάσαμε την τεκμηρίωση που υπέβαλε ο αναφέρον. Εξετάσαμε τις διαθέσιμες πληροφορίες από τις Ιταλικές Περιβαλλοντικές Αρχές ε, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου περιβάλλοντο Και είδαμε ότι για το έργο αυτό. Ε, έχει εκπονηθεί πλήρης ε, μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, που εκπονήθηκε από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι τον Ιούλιο του 2017 με πολλές επιπλέον αξιολογήσεις, επιπλέον έγγραφα, παρατηρήσεις του κοινού, εμπειρογνωμόνων, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όλα αυτά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, αυτής της αξιολόγησης, ήταν ε, η υιοθέτηση διατάγματος ε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος ε, στις 25 Ιουλίου του 2017, που έδειχνε την περιβαλλοντική συμβατότητα του έργου αυτού ε, σύμφωνα με μια σειρά ε, στοιχεία που αναφέρονται στο διάταγμα. Δεδομένου ότι έχει υπάρξει πλήρης ε, μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου για το έργο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνει να έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Όσον αφορά τις ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα που έθιξαν οι αναφέροντες, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι αυτά τα θέματα ήδη καλύπτονται σε δύο διαφορετικές διαδικασίες επιπαραβάση για την παραβίαση των οριακών τιμών ε, της οδηγίας 2008 κάθετο 50 ΕΚ για παραβιάσεις που συνεχίζονται. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε σε τι φάση βρίσκονται αυτές οι διαδικασίες επί παραβάση. Το γνωρίζουμε αυτό. Ξέρω ότι είναι ευαίσθητο θέμα, αλλά αν έχετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία, αυτή τη στιγμή έχει σταλεί μια εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση στις Ιταλικές Αρχές. πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία, διότι ε, εφόσον γνωρίζει η Επιτροπή μας ε, ότι υπάρχει ανοιχτή διαδικασία επί παραβάση, είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε σε τι φάση βρίσκεται η διαδικασία αυτή. Ε, δίνω το λόγο τώρα στους Ευρωβουλευτές. Η κυρία Εύη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που κατέθεσαν την αναφορά που είναι μαζί μας σήμερα. Είναι σημαντικότατη η αναφορά αυτή. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο το οποίο παρουσίασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχουν παραβιάσεις από πλευράς, πιθανές παραβιάσεις από πλευράς της Ιταλικής Διοίκησης και τώρα βρισκόμαστε στην φάση της αιτιολογημένης γνωμοδότησης σε σχέση με την παρουσία του οξυδίου του αζότου και σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Αυτό το οποίο με εκπλήσει όμως, θα ήθελα να πω στα πλαίσια της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ότι στο εσωτερικό των προβλέψεων της υπουργικής απόφασης υπάρχουν 200 περιβαλλοντικές παρατηρήσεις οι οποίες θα ζητηθούν επίσης και από τους Δήμους και τις κοινότητες της περιοχής που δεν έχουν και τα μέσα για να τα παρακολουθήσουν όλα αυτά. Το βασικό είναι ο συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση της κατάστασης, της ποιότητας του αέρα. Η Ιταλία βρίσκεται στην αρχική φάση εφαρμογής ε, των διαδικασιών ελέγχου ε, της ποιότητας του αέρα. Ε, υπάρχει έλλειψη ουσιαστικά μέσων παρακολούθησης της κατάστασης και αναρωτιέμαι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανησυχεί γι' αυτό. Από τη μία ζητάτε από την Ιταλία να παρακολουθήσει την κατάσταση και από την άλλη έχει πολύ λίγες μονάδες παρακολούθησης που έτσι κι αλλιώς δίνουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι ανώτατα, τα ανώτατα όρια δεν γίνονται σεβαστά. Αυτό δημιουργεί δυσφορία και δημιουργεί και οργή από πλευράς συναδέλφων απέναντι σε αυτούς τους τσιμεντένιους γίγαντες που θα παραβιάσουν το έδαφος των περιοχών τους και θα βλάψουν ένα οικοσύστημα που θα έπρεπε να προστατεύεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και αναφέρομαι στην οδηγία Χάμπιτα, όπως επίσης και στην οδηγία για τα πτηνά. Ταυτόχρονα θέλω να διευκρινίσω σχετικά με την οδηγία το ότι οι τοπικές αρχές έχουν ζητηθεί να υπάρξει μια περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων για δύο διαφορετικές περιοχές περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ζώνες ειδική ε, προσοχής και παρατήρησης. Συνεπώς ε, υπήρξαν δύο γνωμοδοτήσεις ταυτόσιμες, ιδιαίτερα επιφανειακές και επιπόλαιες στην ανάλυση τους. Είναι λοιπόν προφανές εδώ ότι πιθανώς ε, θα υπάρξει βλάβη εις βάρος της χλωρίδας και της πανίδας συνολικά. Συνεπώς λοιπόν η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε από το Ιταλικό κράτος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης ήταν ανεπαρκής. Σε πολιτικό επίπεδο θα ήθελα να πω ότι αυτό το σχέδιο δεν είναι α, χρήσιμο για τους πολίτες δεν επιλύει τα προβλήματα κινητικότητας και δεν καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο το οποίο είναι ξεπερασμένο, παλαιό, δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. Και σίγουρα δεν θα μειώσει αν θέλετε την ατμοσφαιρική μόλυνση δυστυχώς ε, αγνοώντας ουσιαστικά όλα τα επιμέρους τοπικά σχέδια προσταχίας ε, της ε, περιοχής που είναι η Βόρεια Ιταλία, η νότια περιοχή του Πάδου που δυστυχώς έχει από τα υψηλότατα επίπεδα θανάτων πρόωρων λόγω της ατμοσφαιρικής μόλυνσης. Είναι δυστυχώς μια θλιβερή πρώτη θέση αυτή την οποία κατέχουμε στην Ευρώπη. Συνεπώς ζητώ την υποστήριξη παρακαλώ των συναδέλφων. Ε, ζητώ να αποσταλούν επιστολές και στις περιφερειακές αρχές ε, για να υπογραμμίσουμε τις ελλείψεις που υπογράμμισαν με τη σειρά τους και αυτοί που κατέθεσαν την αναφορά και να καταγγείλουμε την κατάσταση και στις αρμόδιες αρχές που δεν έκαναν αυτά τα οποία περιμένουν οι πολίτες. Οι Ιταλικές αρχές αγνόησαν τους πολίτες και τα προγράμματα αυτά επαναλαμβάνω είναι άχρηστα και αναχρονιστικά. Ευχαριστώ η κυρία Βαλίνα. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για τις παρουσιάσεις τους και να πω ότι τους υποστηρίζουμε. Πιστεύω ότι δυστυχώς είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες βλέπουμε ε, να μην εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικές οδηγίες και κυρίως επιπλέον ε, υπάρχουν πάρα πολλά προσκάωματα τα οποία δημιουργούν τα ίδια τα κράτη-μέλη για να μην επιτρέπουν την σωστή εφαρμογή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εγώ νομίζω ότι εδώ και ήδη ακούστηκε πρόκειται για ένα έργο το οποίο ε, έχει ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια και είχε μια αντίστοιχη πορεία και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και στις Ιταλικές αρχές ότι το να ε, κατακαιρματίσουμε τις ε, διαδρομές αυτές ε, είναι ε, παραβίαση των περιβαλλοντικών οδηγιών. Πρέπει να γίνει κατάλληλη λοιπόν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρέπει να έχουμε και σωρευτικά μελέτη όλου του αντικτύπου. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία σίγουρα θα πληγεί από αυτό το έργο εάν συνεχίσει η κατασκευή του. Γι' αυτό ακριβώ και πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τι μοντέλο γεωργίας θέλουμε για να μπορέσουμε να ε, προσεργήσουμε από εδώ μέσω της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής ε, την κατάλληλη ασφάλεια τροφίμων που πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον αντίκτυπο του έργου νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε να, ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανεξάρτητη και αυτό είναι πολύ σημαντικό και επικαιροποιημένη και πρέπει να γίνει και μια δημόσια διαβούλευση, κάτι το οποίο από ό,τι ακούσαμε δεν έγινε, για να γίνει σεβαστό τα όσα προβλέπονται από τη σύμβαση του Άρχους. Ε, και θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει λοιπόν ανοιχτή αναφορά και η Επιτροπή μας είπε ότι ήδη θα στείλει επιστολή στις Ιταλικές Αρχές και νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και εμείς ε, ε, να μας διασκεδάσουν τις ανησυχίες μας οι Ιταλικές Αρχές κυρίως όσον αφορά την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και επίση, η Επιτροπή θα πρέπει να μα διευκρινίσει αν υπάρχει χρηματοδότηση, αν προβλέπεται χρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση στο έργο και αν όντω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αν πράγματι υπάρχουν ε, ευρωπαϊκά κονδύλια, τότε σίγουρα θα πρέπει να στείλουμε και επιστολή στην Επιτροπή περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί όχι και στην ε, Επιτροπή περιβάλλοντο για να γνωμοδοτήσουν και αυτοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεται δεν θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φεριόλη λοιπόν και μετά στον κύριο Ταλιαβιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα είπατε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για μας. και ήθελα να επισημάνω επίσης ότι το προηγούμενο έργο για τον αυτοκινητόδρομο ήταν ένα έργο το οποίο ε, άρμοζε πλήρως στην κατάσταση. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε και μετά διεκόπη. Έχουν κατασκευαστεί ελάχιστα χιλιόμετρα και σταματούν πουθενά, στο πουθενά, σε ένα διέξοδο. Επειδή λοιπόν το έργο αυτό ε, θα στοιχήσει το 1 πέμπτο από ό,τι θα στοιχήσει αυτός ο αυτοκινητόδρομος και αρκεί ε, γιατί πρέπει να καταστρέψουμε μια περιοχή όταν υπάρχει ήδη λύση και μάλιστα ε, υπάρχει και δίπλα σιδηρόδρομος και η Ευρώπη βλέπει με θετικό μάτι την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών δικτύων. Πραγματικά ελπίζω η Επιτροπή σας να καταφέρει να αποστείλει ένα σαφές μήνυμα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και στις ε, περιφερειακές αρχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Σταλιαβιάννη. Ευχαριστώ. Δύο σχόλια μόνο και θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Φεριόλη. Το έργο αυτό καταγγέλλεται διότι καταρχάς από οικονομική σκοπιά, πέραν του κόστους που είναι τεράστιο, δεν μας δόθηκε ποτέ μια αποδεδειγμένη, τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ότι αυτό το έργο μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, όπως μας λένε. Δεύτερον, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία κυρίως βασίζεται στην ποιότητα. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς η ποιότητα πρέπει να μεταφέρεται μέσω αυτοκινητοδρόμου όταν υπάρχουν μέσα τα οποία μπορούν να ε, καλύψουν και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό όλες αυτές τις ανάγκες. Ε, δεύτερον, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μια τεχνική επιτροπή η οποία ανέφερε ότι ε, εκμεταλλευτήκαμε όλες τις ε, απαραίτητες οδούς. Η ερώτηση ενός πολίτη, όχι ενός εμπειρογνώμονα, είναι πώς είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι εκμεταλλευτήκαμε όλες τις πιθανές οδούς με κατάλληλο τρόπο, ε, με τυπικό τρόπο, όταν υπάρχουν πάνω από 200 αναλύσεις, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ένα έργο θα πρέπει τουλάχιστον να προσαρμοστεί ε, σε αυτές τις ε, παρατηρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος ώστε να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι παρατηρήσεις στο έργο και μετά θα τα ξανασυζητήσουμε. Διότι και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν επακριβώς τι θα κατασκευαστεί. Ευχαριστώ. Fine. Um, Λοιπόν σα ζητώ να κλείσετε παρακαλώ, δεν είναι εύκολο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι έχει εξαντλήσει τις δυνατότητε. και ότι δεν υπάρχει παραβίαση ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά εσείς συνεχίζετε να ανησυχείτε και συνεπώς και εμείς ανησυχούμε. Ε, νομίζω ότι θα κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή και θα στείλουμε μία επιστολή στις αρχές της Εμίλια Ρωμάνια διευκρινίζοντας ότι πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή η οποία λέει όποιος μολύνει πληρώνει και θα πρέπει να ανησυχήσουν οι αρχές για την ευημερία και την υγεία των κατοίκων της περιοχής και να αναφερθούμε φυσικά στις ε, διαδικασίες επί ε, παραβάση οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στις διαδικασίες αυτές, αλλά πρέπει να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας και να τονίσουμε επίσης ότι γενικά δεν είμαστε καθόλου ε, υπέρ παραβιάσεων κανόνων και ρυθμίσεων. Λοιπόν, ναι μεν η Επιτροπή έχει εξαντλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στάδια, αλλά νομίζω ότι οι ανησυχίες παραμένει. Θα πρέπει να δούμε αν πράγματι το θέμα αυτό έχει καλυφθεί και εμπλέκονται και ευρωπαϊκά χρήματα. Οπότε να δούμε τι γίνεται με τις παρατηρήσεις αυτές και τις πιθανές παραβιάσεις. Μήπως θα πρέπει να ζητηθούν πίσω τα χρήματα τα κοινοτικά, μήπως θα πρέπει να σταματήσει η χορήγησή τους. Ναι, το ξέχασα και αυτό λέει η Πρόεδρος. Θα στείλουμε και μια επιστολή στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων για τις πιθανές ε, παραβιάσεις και για τον τρόπο με τον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί ίσως καταχρηστικό τρόπο οι ευρωπαϊκές πιστώσεις. Παρακαλώ κλείνουμε προς το παρόν την συζήτηση εδώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και παρουσιάσατε με σωστό τρόπο την υπόθεσή σας. Τώρα περνάμε ε, στο Νο Ταντζεντσιάλε, Πάρκο Ντελτιτσίνο. Υπάρχουν πάρα πολλές υπογραφές ε, εναντίον της δημιουργίας ενός πυκνού δικτύου οδικών υποδομών. Έχουμε αρκετούς, ε, τέσσερις. Θα δώσω το λόγο από δύο λεπτά στον καθένα. Θα ξεκινήσω με την Ανιέζε Γκουερέσκη. Χαίρομαι που κάθομαι δίπλα σε Ιταλό και με διορθώνει, λέει η Θα κάνω λιγότερα λάθη από ό,τι στο παρελθόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας που ε, συμφώνησε να συζητήσει την αναφορά μας. Εδώ και 16 χρόνια παρουσιάστηκε ένα σχέδιο δρόμου μεγάλης ταχύτητας που θα συνέδεε το αεροδρόμιο της Μαλπένσα με το δυτικό περιφερειακό οδικό δίκτυο ε, του Μιλάνου. Θα πέρναγε μέσα από το Εθνικό Πάρκο του Τιτσίνο που είναι αναγνωρισμένο σαν πεδίο υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Το 2015 υπήρξε τροποποίηση του σχεδίου αυτού, ακυρώθηκε η σύνδεση με το περιφερειακό και υπήρξε πρόβλεψη σύνδεσης με το Βιτζέβανο, μια συγκεκριμένη μικρή πόλη ε, φυσικά μαζεύτηκαν 14.000 υπογραφές εναντίον της σύνδεσης αυτής. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα με την ενίσχυση του υπάρχοντος οδικού δικτύου και με κυρίως την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι 14.000 αυτές των υπογραφών δείχνουν το ενδιαφέρον του τοπικού πληθυσμού ε, προσφύγαμε και στο τοπικό δικαστήριο, οργανώσαμε πάρα πολλές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, η πιο μεγάλη έγινε το 15 στην περιοχή. Όλες οι περιβαλλοντικές Ιταλικές οργανώσεις συμφώνησαν με τα αιτήματά μας. Εμείς θελήσαμε να δείξουμε ότι το νέο τροποποιημένο σχέδιο είναι μεν διαφορετικό από το αρχικό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει άξι αδειοδότησή του με περιβαλλοντικές επιπτώσεις που είχαν καταμετρηθεί για άλλο σχέδιο και 10 χρόνια νωρίτερα. Συνεπώς λοιπόν η άδεια για την κατασκευή δεν πρέπει να θεωρείται ε, ως ισχύουσα. Κανένα πρόγραμμα οδικών υποδομών δεν μπορεί να γίνει δεκτό αγνοώντας τους πολίτες της περιοχής και γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι μόνο με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της περιοχής μπορούμε να καταλήξουμε σε προγράμματα κινητικότητας που καλύπτουν τις ανάγκες τους, που είναι συμβατά με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής και που σέβονται την βιοπικιλότητα και τις αγροτικές δραστηριότητες στο εσωτερικό αυτών των δύο προστατευομένων περιοχών δεν πρέπει να εμένουν οι αρχές σε αναχρονιστικά προγράμματα. Και έχουμε μαζί μας ένα εκπρόσωπο των γεωργών και δύο δήμαρχους της περιοχής που θα μιλήσουν για τις δικές τους περιοχές. Με πολύ κομψό τρόπο δώσατε το λόγο στους εκλεγμένους πολιτικούς, γιατί συνήθως τους δίνουμε το λόγο και δεν μας τον δίνουν πίσω. Λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί, ας καλωσορίσουμε τους δύο δημάρχους τον κύριο Πιολτίνη και τον κύριο Μπόνα. Τον λόγο ε, έχει ο κύριος Πιολτίνη. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Λέγομαι Τζοβάνι Πιολτίνη, είμαι δήμαρχος της ε, περιοχής του Ολμπαϊράτε 4.300 κατοίκους έχουμε με μεγάλη αγροτική παραγωγή και έχουμε ε, πολλά ύδατα στην περιοχή. Βρισκόμαστε 20 χιλιόμετρα από το Μιλάνο. Ο Δήμος μας ήταν πάντα κατά του συγκεκριμένου έργου γιατί έχει πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Είναι παροχημένο, τεράστιο, πολύ δαπανηρό και σε καμία περίπτωση δεν λύνει τα προβλήματα της τοπικής βιωσιμότητας. Η λύση είναι να υπάρχουν άλλες βιώσιμες παρεμβάσεις χαμηλότερου κόστους και μάλιστα ε, βελτίωση του παρόντος οδικού δικτύου, δυνατότητες επίσης ε, για σιδηροδρόμους και νέο οδικό δίκτυα και ε, ε, ποδηλατοδρόμους μεταξύ των δήμων που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Οι οδικές υποδομές ε, που αμφισβητούμε θα έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες, κυρίως ε, στο Δήμο μας, στο Αλβαϊράτε, που βασίζεται κυρίως ε, στην ομορφιά του τοπίου και στην γεωργία ποιότητας το 42% της επιφάνειας του έργου επιβαρύνει την περιοχή μας και κατά 30% γόνιμες γεωργικές περιοχές. Θα δημιουργήσει ζημίες στο επιφανειακό και στο ε, ε, δίκτυο υδάτων στο υπέδαφο, ε, θα υπάρχουν ζημίε στην επικοινωνία και φυσικά και στη βιοπικιλότητα. Γι' αυτό ακριβώ ζητούμε να διαγραφεί οριστικά αυτό το άχρηστο και δαπανηρό έργο, το οποίο δεν έχει κάνει και κατάλληλη αξιολόγηση κόστου και ωφέλου. Πρόκειται απλώ για τσιμέντο το οποίο επιβάλλεται άνωθεν και δεν λαμβάνει υπόψη του στη σημασία του εδάφους και τι ροέ της κίνησης που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την παρούσα κατάσταση. Επιπλέον, η διαγραφή ε, του έργου θα ε, βελτιώσει την κατάσταση γιατί αλλιώς θα επιδεινωθεί πάρα πολύ η κίνηση στο Δήμο του Αλμπαϊράτε. Τέλος, πρέπει να πω ότι μας εξέπληξε αρνητικά η αλλαγή πορείας για το έργο αυτό από το ε, Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στην Ιταλία στις 27 Ιανουαρίου του 2017 ε, παρέπεμψε στο Άνας ε, το έργο και είπε ότι δεν συμμορφώνεται με την νομοθεσία και πρέπει να υπάρχουν ε, ε, πολύ σημαντικές και ουσιαστικές ε, ε, αλλαγές. Αντίθετα όμως, στην επόμενη συνεδρίαση ενέκρινε το έργο αυτό με κάποιες παρατηρήσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει εντελώς την προηγούμενη γνωμοδότηση. Κατά την άποψή μας η διαδικασία αυτή δεν είναι σύνομη και αυτή τη στιγμή γίνεται και κάποια νομική μελέτη επί του θέματος. Θα πρέπει να λάβει υπόψη τους κάποιες προσθήκες και να λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοκρατίας δημοσίων έργων που εκφράστηκε στις 27 Ιανουαρίου. Ανταυτού, μετά από την προβολή ε, στην αρμόδια επιτροπή, ε, αποφασίστηκε να γνωμοδοτήσει, χωρίς όμως στη συνέχεια να λάβουμε και να εξεταστούν προληπτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία από την Επιτροπή και ε, υπάρχουν κάποια έγγραφα τα οποία ακόμα και σήμερα 11 Οκτωβρίου 2017 δεν έχουμε λάβει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Χίλια ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Ο κύριος Μπόνα, ο δήμαρχος της Καζινέτα Ντιλουγκανιάνου. Πολύ ωραία φαίνονται όλα αυτά τα μέρη και έχουν και υπέροχες ονομασίες. Μακάρι να μπορούσα να τις προφέρω και σωστά. Αν θέλετε μπορείτε κάλλιστα να έρθετε να δείτε την πόλη μας ευπρόσδεκτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δίδετε την δυνατότητα να είμαστε μαζί σας σήμερα. Η καζινέτα τη Λουγκανιάνο ήδη από το 2007 έχει ζητήσει να σταματήσουν τέτοιου είδους έργα και εμείς είπαμε ότι δεν έχουμε περιθώρια περαιτέρω οικοδόμησης και κάλυψης του εδάφους ιδιαίτερα στα πλαίσια του Εθνικού Πάρκου του Τιτσίνο, στο οποίο ανήκουμε. Και αυτό είναι απαραίτητο και ε, για να διασώσουμε τον τελευταίο πράσινο πνεύμονα της κοιλάδας του Πάδου στο νότιο τμήμα της πόλης του Μιλάνου. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, επίσης ε, επιχειρήσεις γεωργικές όπου καλλιεργούνται βιολογικά προϊόντα, 11 είδη βιολογικών αρχαίου τύπου σιτηρών. Ε, ένας δρόμος σαν και αυτόν δεν θα οδηγήσει στο Μιλάνο πια, έχει καταργηθεί η σύνδεση με τον περιφερειακό της πόλης, θα είναι μια άχρηστη λωρίδα ασφάλτου που θα πληγώνει το νότο της Λομβαρδίας, ε, κάτι το οποίο θα καταβροχθήσει τις γεωργικές περιοχές 8 τετραγωνικά μέτρα αναδευτερόλεπτο απώλειας καλλιεργούμενου εδάφους. Ζητάμε βοήθεια από την Ευρώπη. Οι λύσεις για την μετακίνηση οδικά προς το Μιλάνο υπάρχουν. Πρέπει να ε, επενδύσουν ελάχιστο τμήμα των 220 εκατομμυρίων που προβλέπονται για το συγκεκριμένο έργο. Θυμίζω ότι η σιδηροδρομική σύνδεση είναι μονής κατεύθυνσης ε, και ταυτόχρονα ε, δεν γίνονται επενδύσεις στα σύγχρονα σιδηροδρομικά δίκτυα τα οποία έχουν οι υπόλοιπες ε, πόλεις της Ευρώπης. Φοβάμαι ότι η απώλεια εδάφους αν δεν δράσετε θα συνεχίσει να καταβροχθίζει τα εδάφη μας και δεν θα μπορέσουμε να κληρονομήσουμε ε, το έδαφος μας στα παιδιά μας. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ και τις ωραίες εικόνες. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ολιβέρο Ντάριο, ο οποίος εκπροσωπεί τους γεωργούς της περιοχής. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Θα ήθελα να προσπαθήσετε να δείτε από πού θα περάσει η σουπερστράντα αυτή, ο δρόμος υψηλής ταχύτητας. Εμείς έχουμε μία από τις πιο προστατευόμενες περιοχές της περιοχής του Μιλάνο. Αποτελείται από δύο τμήματα, το πάρκο του Τιτσίνο, το Εθνικό Πάρκο και το Εθνικό Πάρκο της Κοιλάδας του Πάδου νότια του Μιλάνου. Νομίζω ότι όπως είπα είμαστε ο πράσινος πνεύμονας της περιοχής μέσα σε μια περιοχή ευρύτερα στο Μιλάνο που είναι από τις πιο μολυσμένες στην Ευρώπη και πρέπει να διευρυνθούν οι περιοχές αντιδικοί μας και όχι να συμπτύσσονται. Θα τροποποιηθεί επίσης το τοπίο των μικρών καναλιών του Μιλάνο κάτι το οποίο είναι παλαιότατο και ε, έχει χαρακτηριστεί και από την UNESCO κάτι το οποίο πρέπει να συντηρηθεί για λόγους πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς. Συνεπώς λοιπόν θα υπάρξουν ε, βλάβες και στο σύστημα των υδάτινων πόρων και κυρίως θα βλάψουν και την παραγωγική μας γεωργική διαδικασία η οποία έχει καταστήσει θα έλεγα την γεωργική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος σαν κάτι το οποίο έχει και οικονομική σημασία και νόημα. Συνεπώς λοιπόν πρόσφατα έχουν δημιουργηθεί και νέες ενώσεις παραγωγών, ενώσεις ε, ε, αυτών που εκμεταλλεύονται ε, σε επίπεδο δασοκομείας τα δάση της περιοχής και υπάρχουν και 30 γεωργικές επιχειρήσεις που παράγουν βιολογικά προϊόντα. Και τίθεται και το θέμα επίσης της συντήρησης του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής και μάλιστα έχουμε πάρει και βραβεία το 2014 και 2015 από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει απόλυτη ενότητα των κατοίκων και των τοπικών συλλόγων εναντίον του δρόμου αυτού υψηλής ταχύτητας δεν μπορούμε πια να ξοδεύουμε τους βιολογικούς και περιβαλλοντικούς μας πόρους και δεν μπορούν τα προβλήματα κινητικότητας να λύονται με απαράδεκτες και απαρχαιωμένες λύσεις και νομίζω ότι εδώ οι παρατηρήσεις τις οποίες συστηματικά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ιταλία ισχύουν και για μας. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γκασπαρινέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω Ιταλικά από σεβασμό και προς τους αναφέροντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θεωρήθηκε παλιό, χαρακτηρίστηκε παροχημένο και είναι από όλες τις μεριές. Είναι υπό την έννοια που μας υπέδειξαν οι δήμαρχοι που είναι εδώ παρέντες σήμερα, αλλά και από νομική σκοπιάς ε, δυστυχώς και εδώ θα πρέπει ε, να δούμε και τη μη αναδρομικότητα της νέας οδηγίας βία. Η αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λάβει και μία ανακοίνωση μέσω της οποίας απαντούμε ε, στα ε, θέματα τα οποία αφορούν το νομικό πλαίσιο όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας βία, η οποία δεν είναι αναδρομική. Πέραν αυτού όμως, αυτή τη στιγμή ε, τέθηκε το θέμα της οδηγίας του 2008 κάθετος 50 και η πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών είχε ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικαιροποιήσει, να ενημερώσει συγγνώμη, τους ε, βουλευτές για αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι μπορώ να σας πω εδώ ότι το συγκεκριμένο έργο μαζί με πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία στην Ιταλία εξακολουθούν να υλοποιούνται παρά το γεγονός ότι υπάρχει κατάφορη παραβίαση της οδηγίας 2008-50 ε, ε, θέτει ένα πρόβλημα το οποίο είναι πλέον και πολιτικό και αυτό πλέον θα πρέπει να το εξελογήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς είναι δυνατόν στην απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη για τις ε, ε, PM10 μας λέει η Ιταλία ότι αυτό θα καλυφθεί το 2025. Το 2025 όταν ε, τα στοιχεία, τα όρια βάση της νομοθεσίας που έχουν εισαχθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δεσμευτικά από το 2005. Υπάρχουν συγκεκριμένε οριακέ τιμέ. Υπήρχε μια πρώτη καταδίκη τη Ιταλία από το δικαστήριο για την ε, ε, παραβίαση των ανωτήτων ε, ορίων του PM, των PM10, των σωματιδίων για το 2007 και το 2008 είναι μια παραβίαση η οποία δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει και επομένως η Ιταλία τίθεται και ενώπιον των ευθυνών τη. Υπάρχουν ελάχιστοι πράσινοι πνεύμονες ε, στη χώρα οι οποίοι θυσιάζονται για ε, παλιές παραχωρήσεις μεταφορών. Πρόκειται απλώ ε, για οικοδομήματα τσιμέντου και δεν είναι η πρώτη φορά που αμφισβητούνται αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός ο πολλαπλασιασμός, ο οποίος δεν έχει και λόγο ύπαρξης. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και οι ίδιοι οι δήμαρχοι μας λένε ότι δεν ανταποκρίνονται στα συμφέροντα της περιοχής. Ε, φοβούμε ε, ότι το πρόβλημα αυτό, όπως και πολλά άλλα προγράμματα υποδομών στην Ιταλία, μπορεί να βρει τη λύση του μόνο στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας επί η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μας φέρει και ενώπιον του δικαστηρίου. Λέω κατά πάσα πιθανότητα, διότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα επισήμως απόφαση και αυτή τη στιγμή σε ένα κράτο μέλο μα απαντά ότι οι οριακέ τιμέ, οι οποίε είναι δεσμευτικέ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το 2005 δεν γίνονται ακόμα σεβαστέ 10 χρόνια μετά και θα αρχίσουν να γίνονται σεβαστέ το 2025 όσον αφορά τη Λομβαρδία και το Βένετο που είναι οι δύο πιο πλούσιε περιοχέ τη Ιταλία. Δεν υπάρχει καν δηλαδή δικαιολογία ε, σαν αυτέ οι οποίε παρουσιάστηκαν από τη Βουλγαρία και την Πολωνία όταν ε, ε, βρέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου και η Βουλγαρία καταδικάστηκε για αντίστοιχα γεγονότα. Υπάρχει λοιπόν προηγούμενη καταδίκη της ε, Βουλγαρίας για την παραβίαση των οριακών τιμών των ε, ορούμενων σωματιδίων. Εάν λοιπόν δεν ληφθεί αυτό υπόψη, θα πρέπει οι Ιταλικές αρχές να λάβουν υπόψη τους όχι μόνο το συγκεκριμένο έργο, ε, το οποίο μπορεί και να είναι και σύνομο με την Ιταλική νομοθεσία. Βεβαίως εσείς μας λέτε ότι υπάρχει ε, προσφυγή ε, στην Επιτροπή ΤΑΡ και σε αυτή τη φάση εφόσον υπάρχει προσφυγή, καλό θα ήταν να περιμένουμε και την απόφαση το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι η προσφυγή στο ΤΑΡ. Υπήρχε και προσφυγή στην Ουνάσκο. Εδώ επιφυλασσόμεθα να απαντήσουμε. Αλλά ε, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η νομοθεσία ούτως ή άλλως ε, έχει οδηγήσει σε μία παραβίαση που έχει τεθεί στο αρχείο. Τώρα, ε, ο νόμος βάσει του οποίου κατασκευάστηκε ο προηγούμενος αυτοκινητόδρομος εξετάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία επί παραβάση ευρωπαικη ενωση η διαδικασια επι ηταν η 2003-3170 αρχιοθετήθηκε και έχει ξεπεραστεί γιατί δεν εφαρμόζονται πια αυτές οι διατάξεις. Ε, επίσης, θα ήταν χρήσιμο εάν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δοθεί και μία πιο σαφής εικόνα όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ του έργου που εγκρίθηκε ε, το 2008 με την βία και την ε, παρούσα εκδοχή. Και σας το ζητώ αυτό, διότι στην αρχική ανακοίνωση προς την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαβάζω ότι αυτή η λειτουργική διαγραφή η οποία αποφασίστηκε και παρουσιάστηκε στους Δήμους το 2015 ως αλλαγή του αυτοκινητοδρόμου, ουσιαστικά ανταποκρίνεται στο προηγούμενο έργο. Εάν όντω ανταποκρίνεται, ο προηγούμενος δρόμος εξακολουθεί να ισχύει. Αλλά από αυτά που άκουσα εγώ σήμερα, κάποιο λέει, η πρώτη παρέμβαση μάλιστα μα το είπε αυτό, ότι το έργο αυτό δεν ανταποκρίνεται με το αρχικό, στο αρχικό. Και επομένως νομίζω ότι μπορώ να διαπιστώσω ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ της γραπτής επικοινωνία που έχουμε ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα όσα ακούσαμε, τον όσων ακούσαμε εδώ σήμερα για το τι ακριβώς συνέβη. Και το πρόβλημα αυτό δεν είναι αδιάφορο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αν αυτό το έργο για το οποίο μιλάμε είναι απλώς ε, η διαγραφή ενός έργου που είχε ήδη εγκριθεί το 2008, όπως λέγεται στην αρχική αναφορά, ή αν πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό όσον αφορά τις νομικές συνέπειες, ε, σαφέστατα υπάρχει διαφορά, διότι μια οδηγία σαν αυτή, η οποία επικαλείστε, που είναι η οδηγία βία, δεν ισχύει αναδρομικά για τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά εάν χρειαστεί να κατασκευαστεί νέος αυτοκινητόδρομος, θα ισχύει η νέα οδηγία. Ζητώ συγγνώμη για την ε, Πρόεδρο, γιατί ε, είναι τόσο νομικά αυτά τα οποία λέω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε κατά πόσον το συγκεκριμένο έργο είναι σύνομο ή όχι και είναι ίδιο με αυτό το οποίο εγκρίθηκε το 2008 γιατί οι νομικές συνέπειες είναι τελείως διαφορετικές. Έχουμε εφαρμογή της νέας οδηγίας. Αυτή είναι απλώς μια αμφιβολία. Ε, αυτό το αφήνω γιατί δεν είναι δική μου δουλειά να διασκεδάσει αμφιβολίες. Αυτό πρέπει να το κάνει αυτός ο οποίος υπέβαλε την αναφορά. Όσον αφορά όμως το γενικότερο πρόβλημα ε, τσιμεντόδρομων αυτών που πραγματικά δημιουργούν προβλήματα στην Ιταλία και όσον αφορά την ποιότητα του αέρα να σας παραπέμψω στην απόφαση που θα πρέπει να λάβει η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι δεν τηρούνται τα ανώτατα όρια των αιρούμενων σωματιδίων και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι παραβιάσεις, εμένουν και βάλουν την Ιταλία στην τρίτη θέση στην Ευρώπη μετά από τη Βουλγαρία και την Πολωνία ε, όσον αφορά τις ημέρες στις οποίες ξεπερνούνται τα ανώτατα όρια αιρούμενων σωματιδίων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμα αυτά που ακούσαμε. Θα σας ζητήσω λοιπόν να μας υποβάλλετε γραπτός τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα είναι πολύ χρήσιμο να τις λάβουμε. Καθότι προσθέτουν ε, νέα στοιχεία σε σχέση με τις προηγούμενες επαφές που είχαμε. Το λόγο έχουν οι ευρωβουλευτές. Ελεονόρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ξεκινώντας θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά αυτούς που κατέθεσαν την αναφορά, τους δημάρχους, τους συλλόγους, τους πολίτες, τους γεωργούς που κινητοποιήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια και έφτασαν εδώ και να ευχαριστήσω επίσης για την πληρέστατη παρουσίαση και απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σαφές ότι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έθεσε τα στοιχεία που θεωρούμε εμείς καθοριστικά, όχι αυστηρά σε νομικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή συμμόρφωσης και εφαρμογής των νομικών ρυθμίσεων, αλλά και σε επίπεδο πολιτικό το οποίο <coughs> εμείς εδώ θα συγγνώμη να εκπροσωπήσουμε. Εδώ και δύο χρόνια είχα πάρει μέρος στην τελευταία κινητοποίηση που είχε γίνει στην περιοχή εναντίον ε, της ε, προσπάθειας αυτής αλλίωσης του περιβάλλοντος και πρέπει να το επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα παράλογο σχέδιο είναι κάτι το οποίο βασίζεται σε απαράδεκτες και ξεπερασμένες αντιλήψεις μια σύνδεση με το αεροδρόμιο της Μαλπένσα που δεν είναι το hub το οποίο επιθυμούσαμε εδώ και 20 χρόνια δεν θα λύσει τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής και τα ειδικά χαρακτηριστικά της. Και δεν θα βοηθήσει και την επικοινωνία της περιοχής αυτής με το κέντρο της πόλης του Μιλάνο. Συνεπώς λοιπόν δεν έχει νόημα και δεν έχει λογική μία τέτοια θα έλεγα κατασκευή και στα εδάφη αυτά δημιουργούνται νέες πραγματικότητες βιολογικής και οργανικής μετάβασης που θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια διαφορετική γεωργία. Υπάρχουν προγράμματα προς την βιολογική παραγωγή ε, προς την προστασία και τον συνδυασμό του περιβάλλοντος και της γεωργίας και δεν πρέπει να απειλούμε τις ε, ενέργειες αυτές. Ε, η περιοχή συνολικά αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα στον τομέα της μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Πρέπει να μην στηρίζουμε την χρήση των ιδιωτικών οχημάτων είναι πολιτική επιλογή να υποστηρίξουμε την συλλογική μετακίνηση μέσα από τα δημόσια μέσα μεταφοράς όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο είναι απολύτως ακατάλληλο, δεν έχει αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε και όμως η περιφέρεια της Λομπαρδία ξοδεύει ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού της ε, στην κατασκευή των οδικών υποδομών και ελάχιστες επενδύσεις κάνει στο σιδηροδρομικό κομμάτι. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα παλαιότυπου. τύπου, οι αξιολογήσεις οι περιβαλλοντικές είναι ξεπερασμένες, δεν είναι σωστή η λογική πίσω από το πρόγραμμα αυτό και απλά ένα τμήμα, μια ένα κομμάτι του προγράμματος αυτού στην ουσία καταστρέφει και τις υπάρχουσες υποδομές και πρέπει να επαναξιολογηθούν οι, ε, τα σχέδια των εργολάβων και σε επίπεδο περιβαλλοντικό. Εμείς λοιπόν σαν τον κίνημα των πέντε αστέρων ζητάμε από την πρόεδρο της Επιτροπής μας να αποστείλει στις τοπικές και εθνικές και περιφερειακές αρχές μια επιστολή ζητώντας τους να ακούσουν τις ανησυχίες των πολιτών διότι είναι απαράδεκτα τέτοιου είδους σχέδια και πρέπει να υπάρξουν λύσεις εναλλακτικές και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις οι οποίες δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη. Αλλιώς να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Η Άντζελα Βαλίνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα προηγούμενα. Καταρχάς αναφερόμαστε στις παγίδες που υπάρχουν για να θεμελιώσουμε αυτά τα εμπόρια τσιμέντου που γίνεται στην πραγματικότητα και είδαμε και τις φωτογραφίες που δεν χρειάζεται, μιλούν από μόνες του. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας διευκρίνησε πάρα πολύ καλά τα πράγματα και μίλησε πολύ σαφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Αυτά τα οποία βιώνουμε ε, τα είπε και ο αναφέρον προηγουμένως. Ε, να δούμε λοιπόν αν εδώ μπορούμε να πούμε ότι ε, αυτό που είπε προηγουμένως και ο αναφέρον, όποιος ρηπαίνει πληρώνει, αλλά αυτός που πληρώνει δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί και να ρηπαίνει. Και πρέπει να δου, πούμε και στην Ιταλική κυβέρνηση πώς πρέπει να πράγματα. Βλέπουμε συνεχώς την παραβίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το βλέπουμε πουθενά και στην περιοχή μου, στη Λαπάλμα και επειδή ε, δεν τηρείται καθόλου και η σύμβαση του Άρχους ε, είναι κατάφορες αυτές οι παραβιάσεις και εδώ επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν και περιφερειακά κονδύλια επομένως ε, πρέπει να τα διαβάσουμε όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι και πολύ αυστηρές οι κυρώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάλλη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι κάτοικος του Μιλάνου 500 μέτρα από το σπίτι μου υπάρχει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ογκολογικό νοσοκομείο που ασχολείται με νεοπλασίες ε, διότι στην περιοχή μου και στο Μιλάνο και στην ε, Λομβαρδία ε, είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει μεγάλη κυκλοφορία ανέμων, δεν υπάρχουν ρεύματα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρήπανση και επομένως κατά συνέπεια ο κόσμος νοσεί. Αυτό φυσικά σημαίνει και αυξημένο κόστος για το Ιταλικό κράτος, διότι προσπαθεί να θεραπεύσει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι βέβαια τις περισσότερες φορές αρρωστώνουν από ανίατες ασθένειες και επομένως ε, έχουμε και πάρα πολλά έξοδα και από πλευρά δημόσια υγεία. Αυτά τα έργα λοιπόν, τα οποία δεν σχετίζονται μόνο με το συγκεκριμένο έργο, αλλά και με πολλά άλλα, είναι αποτυχία προγραμματισμού και για την κοινωνία μα, αλλά και για την περιοχή μου ε, πιο συγκεκριμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη μα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επαληθεύσουμε και από περιβαλλοντική σκοπιά κατά πόσον ε, είναι παροχήμένε αυτέ οι μελέτε και από οικονομική σκοπιά, διότι πολύ συχνά μου έχει συμβεί να βλέπω τέτοια έργα τα οποία όλα βασίζονται σε εκτιμήσεις κυκλοφοριακής κίνησης οχημάτων, ε, τα οποία όμως δεν οδηγούν και σε αποζημίωση για την επένδυση. Υπάρχει, για παράδειγμα, παράδειγμα της ε, ε, Ανατολικής Τανσενσιάλε αντίστοιχα έργα στα οποία υπάρχει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, έχει συμβάλει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μετά επειδή είναι δημόσια η εγγύηση, οι τελευταίοι, ε, ε, οι τράπεζες οι οποίες θα έπρεπε να δίνουν κάτι για αυτές τις επενδύσεις δεν είναι αυτοί που πληρώνουν αλλά επιβαρύνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα οι ευρωπαϊκές δομές θα πρέπει να προστατεύσουν τους πολίτες στην περιοχή μου για να αποφύγουμε ε, από τις πολιτικές οι οποίες οδηγούν στη διαχείριση των ε, μειοδοτικών διαγωνισμών, στις οποίες ε, πολύ συχνά εμπλέκεται και η μαφία στη χώρα μου, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει, διότι πραγματικά έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και όσον αφορά τη ρήπανση και τη διαχείριση των ε, κονδυλίων και την υγιή διαπάνη λοιπόν των δημοσίων κονδυλίων και είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει αυτή η αναφορά ανοιχτή για να πιέσουμε ώστε οι επιλογές του δημοσίου να είναι πιο ε, σοβαρές σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους ε, συναδέρφους που ήταν σχετικά σύντομοι. Ε, να στροφώ και πάλι στον αναφέροντα ε, για να μας ε, κάνετε μια πολύ σύντομη παρέμβαση με βάση αυτά που μόλις ακούσατε. Λοιπόν, η σύνδεση της Μαλπένσα με την, με τον περιφερειακό, το δυτικό κομμάτι του περιφερειακού του Μιλάνου είναι κάτι το οποίο εκρεμεί. Ε, έχει θεωρηθεί ε, κάτι το δευτερεύον ενώ αυτό δεν είναι σωστό και ταυτόχρονα η σύνδεση με το Βιτζέβανο είναι και αυτή κάτι το δευτερεύον σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό. Ο δρόμος αυτός δεν μπορεί να είναι ε, αυτό το οποίο προβλέπεται, ένας δρόμος δηλαδή με πάρα πολλές διακοπές, ένας δρόμος ο οποίος δεν καταλήγει στον περιφερειακό, ένας δρόμος ο οποίος δεν εξυπηρετεί την κινητικότητα των κατοίκων. κανονικά θα έπρεπε να έχουν σαν στόχο το Μιλάνο και όχι το αεροδρόμιο της Μαλπένσα, κάτι το οποίο αποτελεί δευτερεύοντα στόχο. Πρόκειται λοιπόν για ένα σχέδιο το οποίο δυστυχώς ε, δεν θα βοηθήσει σε τίποτα και μάλιστα η κατασκευή τμηματική αυτού του δρόμου θα δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα, θα φέρει στην περιοχή ένα τμήμα της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και στην ουσία θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει. Το σχέδιο το τελευταίο που κατατέθηκε το 2015 επαναλαμβάνω δεν είναι σωστό. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έγινε αμέσως μετά παραπέμπει στην παλαιότερη μελέτη αλλά δεν, είναι, δεν πρόκειται για το ίδιο σχέδιο ουσιαστικά οπότε δεν ισχύει η μελέτη αυτή. Να προσθέσω εδώ επίσης ότι το σχέδιο αυτό μας ε, επιβάλλεται. Στην ουσία ε, είναι κάτι το οποίο μας λένε δεν μπορείτε να το αποφύγετε είναι κάτι το οποίο αποφασίστηκε και δεν μπορείτε εσείς να το αλλάξετε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ξοδέψει χιλιάδες χρήματα για τις μελέτες και δεν μπορεί να αλλάξει τώρα πια. Αλλά δεν πρέπει να ισχύσει αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Νομίζω ότι υπάρχει γενική συνένεση ότι χρειάζεται να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να στείλουμε επιστολή στην, ε, στο, στα Υπουργεία ε, Περιβάλλοντος Υποδομών ε, Μεταφορών καθώς και στις τοπικές αρχές της Ιταλίας και να τονίσουμε την σημασία της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και να τους καλέσουμε να συνεχίσουν τον διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι νιώθω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι με το μέρος μας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία χρειάζεστε, χρειάζεται να υποβάλλετε εσείς οι αναφέροντες ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν ε, είχαν συμπεριληφθεί αρχικά. Σας καλώ λοιπόν να συνομιλήσετε μεταξύ σας ε, εγκαταλείποντας την αίθουσα και να δώσετε τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αντίγραφο προς την Επιτροπή Αναφορών. Έτσι θα λάβουμε και εμείς επικαιροποιημένες τις πληροφορίες ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γραπτός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι τις Βρυξέλλες. Ε, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά και θα συνεχίσουμε να, να παρακολουθούμε την κατάσταση διότι είναι τόσο όμορφο αυτό το μέρος της Ευρώπης. Ε, θα είναι κρίμα να καταστραφεί. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιστροφή σε αυτήν την όμορφη γωνιά της Ευρώπης. Να απευθυνθώ στον κύριο Μαριά που είναι ε, εισηγητής ε, σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής ε, Αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 216 του κανονισμού της εργασίας της Επιτροπής μας κατά το έτος του 2016. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία στενής συνεργασίας ανάμεσα στον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές ε, για να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε την έκθεση αυτή μέχρι το τέλος της χρονιάς, διότι είναι τόσο σημαντική αυτή η έκθεση. Κύριε Μαριά. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για τη συνεργασία που είχαμε, για την προσπάθεια να συγκροτηθεί αυτή και η πρόταση ψηφίσματος ουσιαστικά και η έκθεση μια έκθεση σημαντική για τις εργασίες της ε, δικιάς μας Επιτροπής για το έτος 2016. Επισημάνω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά που είμαι ε, ραπορτέρ σε αυτή την έκθεση. Το 1994 είχα ασχοληθεί ως πανεπιστημιακός δάσκαλος με το δικαίωμα αναφοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα είχα γράψει και επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά. Και χαίρομαι που υπάρχει και αναφορά στο άρθρο μου «The right to petition the European Parliament after Maastricht» το οποίο αναφέρεται και στην μελέτη που έγινε και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πω λοιπόν ότι α, είναι πολύ σημαντικό το δικαίωμα αναφοράς διότι δίνει την ευκαιρία στους πολίτες όπως είδαμε πριν λίγο ε, συμπολίτε μας ε, και φίλους από την Ιταλία να έρχονται εδώ και να θέτουν τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Και είναι η μοναδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία έχουν άμεση παρουσία και συμμετοχή οι πολίτες. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Το είχα τονίσει από το 1994 στα άρθρα που είχα γράψει και μάλιστα αξιοποιώντας την ε, δυνατότητα ε, που μου δίνει η θέση του εισηγητή ε, στη δομή της έκθεσης, στο δεύτερο μέρος υπάρχει ε, η αιτιολογική έκθεση. Και στην αιτιολογική έκθεση ε, παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία για το πώς ασκείται το δικαίωμα αναφοράς, διότι είναι γνωστό ότι στην έκθεση έχουμε περιορισμένο ε, χώρο και αριθμό λέξεων για να ετοιμάσουμε την έκθεση. Αναφέρω λοιπόν ότι το 2016 είχαμε 1569 αναφορές ενώ το 2000 είχαμε μόνο 908 αναφορές που δείχνει ότι υπάρχει μια αύξηση των αναφορών. Όμως είναι λίγες σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ε, συμπολιτών μας. Το δεύτερο θέμα που έχει ενδιαφέρον είναι η ότι περισσότερες αναφορές κρίνονται παραδεκτές 1110 έναντι 450 των μη παραδεκτών το 2016. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι αναφορές, πρωταθλήτρια είναι η Ιταλία, είδαμε και πριν λίγο τους ε, ε, φίλους από την Ιταλία, με δεύτερη τη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι στην 8η θέση ε, που δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών, κυρίως με τα πολλά προβλήματα που έχουν λόγω της πολιτικής που ασκεί η Τρόικα στην πατρίδα μας. Ε, σε επίπεδο γλωσσών, τα αγγλικά είναι η πρώτη γλώσσα που χρησιμοποιούνται από τους αναφέροντες, με τα ιταλικά ως δεύτερη γλώσσα. Τα ελληνικά δεν πάνε άσχημα, είναι στην 8η θέση. Η ηθαγένεια του κράτους μέλους, πάλι έχουμε Ιταλία, ε, Ιταλική ηθαγένεια, Γερμανική ηθαγένεια, Ισπανική και Ελληνική στην 8η θέση. Ε, τα θέματα που μας αφορούν είναι η εσωτερική αγορά, τα θέματα δικαιοσύνης, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η υγεία, κοινωνικές υποθέσεις, απασχόληση, εκπαίδευση και πολιτισμός. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλα τα βασικά θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες έχουν έρθει εδώ. Για την Ελλάδα που έχει ενδιαφέρον και μας παρακολουθούν και αυτή τη στιγμή αρκετοί φίλοι μέσα από το Facebook, διότι κάνουμε live μετάδοση την ε, συζήτηση που γίνεται μέσα από το δικό μας Facebook και, το, και την ιστοσελίδα που έχουμε, κάτι το οποίο κάνουμε συνεχώς ε, απασχόλησαν θέματα όπως είναι το ελληνικό, μια δίθεν επένδυση η οποία απασχολεί αυτή τη στιγμή την Ελλάδα, το θέμα της εξόριξης χρυσού στη Χαλκιδική, το θέμα του χιτά της φυλής όπου τώρα ξαναεπεκτείνεται το χιτά της φυλής, μια απαράδεικτη κατάσταση, θα έρθει καινούργια αναφορά κυρία Πρόεδρε, οι υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών, τα δικαιώματα των μικροομολογιούχων που καταστράφηκαν από το PSI, ε, μέτρα της Τρόικας κατά των δικηγόρων του Αιγείου και το σημαντικό θέμα που έχουμε θέσει κυρία Πρόεδρε και το λέμε και στην έκθεση το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Ένα θέμα το οποίο ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας εκρίθη η αναφορά 22-14 του 2014 των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ως παραδεκτή με παρέμβαση δική μας στις 7 Σεπτεμβρίου του 2015 δυστυχώς οι συντονιστές, η πλειοψηφία των συντονιστών, των συναδέλφων μας στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 ζήτησαν να κλείσει η αναφορά διότι λέει δεν εμπίπτει δήθεν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξήγησα τότε ότι εμπίπτει, διότι είναι ένα σοβαρό θέμα, αφορά τις σχέσεις Ελλάδας με τη Γερμανία, αφορά τη δικαίωση χιλιάδων θυμάτων που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχή αφορά την επιστροφή του κατοχικού δανείου από πλευράς Γερμανίας στην Ελλάδα, ένα θέμα σοβαρό εν ώψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και τα οικονομικά θέματα της Τρόικας Κακώς κατά την άποψή μας κρίθηκε. Αυτό βεβαίως ήταν απόφαση της πλειοψηφίας. Αλλά και αυτό που συνεχίζεται κυρία Πρόεδρε και το είπα και προηγουμένως είναι ότι δεν δέχεται η Επιτροπή μας να κάνει ούτε μία δημόσια ακρόαση για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Απερίφθησαν επανειλημμένα οι προτάσεις μας κάθε χρόνο για το θέμα αυτό και δυστυχώς κυρία Πρόεδρε πριν λίγο όταν συνεδριάζαμε ξανααπερίφθη από όλες τις πολιτικές ομάδες συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς η πρότασή μας να έχουμε δημόσια συζήτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ίσως πλέον η ΓΚΟΕ μου έκανε εντύπωση το ότι καταψήφισε την πρότασή μας για δημόσια συζήτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ίσως θέλει να διευκολύνει την ελληνική κυβέρνηση η οποία δεν προχωρά στο θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων. Ε, στην έκθεσή μας, κυρία Πρόεδρε, αναφερόμαστε στα μεγάλα θέματα τα οποία απασχολούν ε, αυτή τη στιγμή τους Ευρωπαίους πολίτες. Το πρώτο θέμα στο σημείο 6 είναι το πώς εφαρμόζεται ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Διότι πρέπει να εφαρμοστεί. Υπάρχει μια ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περιοριστική. Ε, λέει ότι δεσμεύονται τα κράτη-μέλη από τον χάρτη μόνο στο βαθμό που ε, υπάρχει εφαρμογής στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς θα θέλαμε μια πιο διευρυμένη ερμηνεία. Στο σημείο 7 αναφερόμαστε σε κεντρικό θέμα που μας απασχόλησε και μας απασχολεί ε, και είναι τι θα γίνει με τα δικαιώματα των συμπολιτών μας μετά τον Brexit. Είδαμε ότι είχαμε πολλές αναφορές, συζητήσαμε το θέμα του Brexit. Μας απασχολεί εμάς εδώ τι δικαιώματα θα διατηρήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, μεταξύ των οποίων και 63.000 Έλληνες, οι οποίοι είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι θα γίνει μετά την αποχώρηση, ποια θα είναι τα δικαιώματά τους. Σημαντική ε, δράση της Επιτροπής μας αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με τα άτομα με αναπηρίες. Είναι δεδομένη η συμπαράστασή μα, η παρέμβασή μα, ο αγώνα που κάνει η Επιτροπή Αναφορών, παρέμβασή μας που θέλουμε να εγκριθεί η συνθήκη του Μαρακές που δίνει δικαιώματα στους τυφλούς ε, και θα έλεγα ότι εκεί είναι μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία λαμβάνουμε. Δύο θέματα σημαντικά που μας απασχολούν στο σημείο 15 είναι τα θέματα παιδικής πρόνοιας, η εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν σχέση με γαμικές διαφορές, ε, υπάρχουν πολλές προστριβές μεταξύ πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ε, της γονικής μέρημνας, μερικές φορές έχουμε ακόμη και απαγωγές παιδιών. Το επόμενο θέμα που επίσης μας απασχολεί είναι στο σημείο 10 για τη διασυνοριακή αναγνώριση των υιοθεσιών. Πηγαίνω όσο πιο γρήγορα μπορώ κυρία Πρόεδρε και τελειώνω. Και τέλος έχουμε ένα θέμα σημαντικό που είναι το δικαίωμα πρωτοβουλίας των πολιτών Κάτι που αναφέρουμε στο σημείο 11 που θέλουμε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Να συγχαρούμε επίσης και την ε, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια με την οποία υπάρχει στενή συνεργασία της Επιτροπής μας και νομίζω ότι ε, περιμένω από τους συναδέλφους που σε λίγο θα λάβουν το λόγο για παρατηρήσεις προκειμένου αυτή η έκθεση να εμπλουτιστεί με τις παρατηρήσεις, με τις τροπολογίες ε, και φυσικά θα κάνουμε το παν για να είμαστε μέσα στους χρόνους για να τελειώσουμε αυτή την έκθεση και να ψηφίσουμε ψηφιστεί εγκαίρω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ε, το 2000 ε, π.Χ. Ε, είπε ένας ε, Ρωμαίος ότι θα πρέπει να καταστραφεί, έλεγε κάθε φορά που του έλεγαν κάτι ότι πρέπει ε, να καταστραφεί η καρχιδόνα. Και αναφέρεστε πάντα σε αυτό το αγαπημένο σας θέμα, ό,τι και να συζητάμε. Αυτό είναι μεγάλο επιτεύγμα. Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να μην το πω. Λοιπόν, Έχουμε κάποιους εσκιώδεις εισηγητές εδώ πέρα. Θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση στην Επιτροπή μας στις 22 Νοεμβρίου για να ε, πάει στην Ολομέλεια στην Σύνοδο του Δεκεμβρίου. Thank you very much. I would, I will use Slovak now. Δίνω το λόγο στον Παουλ Τσάκη. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σλοβακικά. Δεν είμαι ε, ο σκιώδης εισηγητής ε, στο θέμα αυτό. Ο κύριος Πρέντα είναι σκιώδης εισηγητής ε, του ΕΛΚ. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκεται σε άλλη επιτροπή και γι' αυτό θα παρουσιάσω εγώ τη θέση του. Ο κύριος Πρέντα επικροτεί την εξαιρετική συνεργασία με τον κύριο Μαριά και Πιστεύουμε ότι ε, ε, το υλικό παρουσιάζεται με πολύ σωστό και επαγγελματικό τρόπο. Ο κύριος Πρέντα τονίζει την ε, αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, την διαφάνεια των αποφάσεων στην Επιτροπή Αναφορών. Η Επιτροπή εργάζεται καλύτερα από τις προηγούμενες θητείες. Και αυτό είναι θετικό για τους ε, συνεργάτες ε, και την ηγεσία της Επιτροπής μας. Ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία βεβαιότητας, δεν ξέρουμε τι συνεπιές θα έχει το Brexit και το ΕΛΚ στηρίζει την ιδέα ότι η Επιτροπή μας αγωνίζεται υπέρ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν και η είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε στο πλευρό των πολιτών. Συμφωνούμε με τον Μαριά σε όλα τα σημεία εκτό από ένα. Γνωρίζετε ποιο είναι αυτό. Είναι το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων προ την Ελλάδα. Ο κύριο Πρέντα ε, λέει ότι το ΕΛΚ δεν θα υπερψηφίσει το σημείο αυτό. και αυτό ισχύει για όλους τους ε, συναδέλφους μας. Ε, εγώ έχω πιο ήπια θέση από τον κύριο Πρέντα, καταλαβαίνω τη θέση του κύριου Μαριά ε, και εκτιμώ τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τα ιδανικά τους. Επιτρέψτε μου προσωπικά να πω κάτι, ότι ο κύριος Μαριάς μου θυμίζει τον πατέρα μου που τη δεκαετία του 1970, πριν 50 χρόνια δηλαδή, επαναλάμβανε ότι πρέπει να πέσει η Σοβιετική Ένωση και ο κομμουνισμός διότι πρόκειται για ανήθικο σύστημα. Το, τη δεκαετία του 70 κανείς δεν το πίστευε αυτό, 20 χρόνια αργότερα όμως ε, πράγματι ε, συνέβη αυτό. Ε, κύριε Μαριά, μπορεί να βρείτε το δίκιο σας σε 20 χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Τζούντ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επικροτήσω και εγώ την έκθεση, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την γραμματεία. Επικροτούμε το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου, θα υποβάλουμε όμως και κάποιες τροπολογίες. Τέσσερα σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Το πρώτο είναι ότι είναι σαφές από τον αριθμό των αναφορών που έχουν υποβληθεί και το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ε, αλλαγή στον αριθμό, ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε ε, όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το δικαίωμά τους ε, να υποβάλουν αναφορές. Θα πρέπει να σκεφτούμε πιο προορατικά πώς θα το κάνουμε αυτό. Ένα ε, τρόπο να γίνει αυτό και εντυπωσιάστηκα από αυτό που είπαν οι αναφέροντε νωρίτερα. Ε, θα πρέπει να δείξουμε λοιπόν πώς ε, έχει λειτουργήσει υπέρ των πολιτών η Επιτροπή μας και πώς έχει πετύχει θετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε καλύτερα πώς οι εργασίες της Επιτροπής μας εντός του Κοινοβουλίου μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις ζωές των πολιτών, μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση και να επιλύσει διαφορές με τη μη δικαστική έννοια. Σημαντικό είναι ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι το μέρος όπου μπορεί να ακουστεί η φωνή των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είναι περίεργο που είχαμε μόνο 61 αναφέροντες παρόντες κατά τη διάρκεια του 2016. Όταν μιλώ εγώ με αναφέροντες έτσι νιώθουν ότι μπορούν να παρουσιάσουν σωστά τις υποθέσεις τους όταν είναι παρόντες και μπορεί να ακουστεί η φωνή τους και μπορούν να συνομιλήσουν απευθείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα. Μπορεί λοιπόν αυτό να ε, μας τρώει πολύ χρόνο, αλλά εγώ θα έδινα προτεραιότητα στο χρόνο που δίνουμε στους αναφέροντές μας. Και όλα αυτά ιδιαίτερα στο πλαίσιο της κρίσης εμπιστοσύνης την οποία έχουμε συζητήσει επανειλημμένα στην Επιτροπή μας. Η ελήφθη η απόφαση το 2016 για την αναφορά που πραγματοποιήθηκε το 2017 στην οποία συμμετείχαμε και οι δύο αλλά ε, είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει πολύ φέτος και η Επιτροπή Αναφορών σαφώς έχει να παίξει ρόλο κλειδί. Πριν ε, το δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, μου έκανε εντύπωση πώς οι πολίτες ε, θεωρούσαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους. Ε, και ε, αναφέρεται το Brexit στην έκθεση, αναφέρεται πολύ σύντομα όμως. Ε, εκείνη όμως τη συγκεκριμένη στιγμή κρίσης, χιλιάδες πολίτες θεώρησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τον τρόπο να μεταφέρουν τις ανησυχίες τους. Και πολλοί ε, πολίτες στην Ευρώπη, 4,5 πολίτες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και στο υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανησυχούν για το τι θα γίνει σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις του Brexit. Και είναι, αξίζει τον κόπο λοιπόν να τονίσουμε αυτήν την παράγραφο για το Brexit στην έκθεση. Καταλαβαίνω πάντως ότι έχει ληφθεί υπόψη και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και δεν το λέω αυτό μόνο επειδή είμαι Ευρωβουλευτής σε Βρετανίδα αλλά ε, αφορά πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφορά όμως και τους Βρετανούς ε, ε, υπηκόους στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικό είναι να τονίσουμε και τις δύο ομάδες πολιτών που θα επηρεαστούν από αυτό. Επίσης, χρήσιμο θα ήταν να βελτιώσουμε την διατύπωση στις απαντήσεις μας για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα εμπιστοσύνης που υπάρχει στην, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο του πληθυσμού. Ε, αναλυτικές και διαφανείς απαντήσεις από την Κομισιόν αλλά και από το Συμβούλιο θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πολύ σπάνια έχουμε κράτη-μέλη να υπερασπίζονται την θέση τους και νομίζω ότι αυτό συχνά είναι εις βάρος της ποιότητας στις συζητήσεις μας. Χρήσιμο θα ήταν για παράδειγμα σε σχέση με τις Ιταλικές αναφορές να είχαμε ακούσει την απάντηση των αρχών. Και τέταρτη παρατήρηση, θα είμαι πολύ σύντομη, το υπόσχομαι. Ε, νομίζω ότι το δίκτυο αναφορών είναι πολύ χρήσιμο. Ανησυχώ λίγο ότι συχνά οι συμμετέχοντες είναι μέλη του, της Επιτροπής μας αλλά που είναι και μέλη άλλων επιτροπών ε, και έτσι δεν ε, διευρύνουμε τον κύκλο ε, και ο Ιάρεκ και εγώ είμαστε μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου έτσι δεν διευρύνεται το δίκτυό μας νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές και το προσωπικό τους σχετικά με το δικαίωμα αναφορών ώστε να ενθαρρύνουν τους πολίτε να υποβάλουν αναφορέ σε αυτούς για να διαδοθεί το μήνυμά μας. Έχει γίνει πολλή δουλειά πάνω στο θέμα αυτό. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Και τελευταία παρατήρηση, νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά ατυχές ε, ο εισηγητή ε, να χρησιμοποιήσει αυτήν την έκθεση για να προωθήσει την δική του εκστρατεία την οποία γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως σημαντική η έκθεση αυτή για τις εργασίες του συνόλου της Επιτροπής. Παρακαλώ λοιπόν να μην διακυβευτεί το σύνολο της έκθεσης ε, για κάτι που έχει ήδη αποφασιστεί σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής μας με δημοκρατικό τρόπο. Αυτή λοιπόν είναι η έκκλησή μου προς τον εισηγητή ε, τώρα που θα προχωρήσουμε στη συζήτηση των συμβασμών. Σας ευχαριστώ πολύ και Φυσικά είναι πολύ ενδιαφέροντες οι συλλογισμοί που μας παρουσιάζετε και είναι χρήσιμο να τα συζητάμε τα θέματα αυτά ε, πότε πότε. Σας ε, καλώ λοιπόν να τροποποιήσετε το κείμενο. Ε, Άντζελα, έχεις το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μαριά για το σχέδιο έκθεσης. Εγώ ήμουν εισηγήτρια πέρσι, ξέρω πως η δουλειά προϋποθέτει και πολύ ευχαρίστω να συνεργαστώ μαζί σας ε, ό,τι χρειαστείτε ως σκιώδης εισηγήτρια βεβαίως. Ε, επειδή αναφερθήκατε στην αριστερά, εγώ θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να ρίξετε μια ματιά στα πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών του 2016 που η αριστερά υπερψήφισε να παραμείνει ανοιχτή αναφορά σας. Υπάρχει μια θετική πλευρά στην αύξηση των αναφυρών, που σημαίνει ότι ναι, μεν υπάρχουν περισσότερα προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και κάτι θετικό, ε, διότι και στον αριθμό των ε, αιτήσεων και στον αριθμό αυτών που κρίνονται παραδεκτές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες γνωρίζουν λίγο καλύτερα αυτό το εργαλείο, γνωρίζουν καλύτερα την Επιτροπή και θεωρούν ότι ε, εμείς τους φροντίζουμε και αναγνωρίζουν και το δικαίωμά τους να υποβάλει αναφορά. Το 2016, όπως επισημαίνει ο εισηγητής, 61 αναφέρονται συμμετείχαν ενεργά στις ε, εργασίες της Επιτροπής. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται, ε, θα μας το διευκρινίσει βέβαια και ο ίδιος, ε, στους αναφέροντες που ήταν παρόντες και που ήρθαν εδώ στην Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοείται. Θα ήθελα να ε, σας συγχαρώ για την έκθεση γιατί από πλευράς της ομάδας μου ε, συμφωνούμε με τα βασικά στοιχεία τα οποία τονίζετε εδώ στην έκθεση. Για παράδειγμα, συμφωνούμε απόλυτα με τα όσα λέτε για την ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών διότι θεωρώ ότι προσφέρει τεράστιες δυνατότητες να ενισχύσουμε ακριβώς αυτή τη συμμετοχή των πολιτών και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή είναι η άποψή μου, εξακολουθεί να θέτει όσο περισσότερα εμπόδια μπορεί ώστε ε, να μην ε, ε, υπάρχουν αποτελέσματα και να διαλύσει τι προσδοκίε των πολιτών που δημιουργήθηκαν αυτή την πρωτοβουλία. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή για τις επικρίσεις ε, προς την ε, περιορισμένη ερμηνεία που δίνεται πάντα στο πεδίο ε, εφαρμογή τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνούμε επίση με την πρόταση για βελτίωση των προθεσμιών και την ποιότητα των απαντήσεων τη Επιτροπή. Είναι ουσιαστικό αυτό. Σήμερα είχαμε ένα παράδειγμα μια εξαιρετική παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ε, εκτέθηκαν σαφέστατα τα πράγματα, και, αλλά υπάρχουν άλλες φορές που δυστυχώς έχουμε δει κάποια παραδείγματα εντελώς αντίθετα και ορισμένες φορές δεν έρχονται και καν, όπως έχει συμβεί σε κάποιες ε, περιπτώσεις και ε, θεωρούμε και πολύ θετική την στενή συνεργασία με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια τίποτα άλλο, να πω ότι υποστηρίζουμε τον προσανατολισμό της έκθεσης και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και με τον εισηγητή και με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες και μέσω τροπολογιών και για ό,τι άλλο χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πει δύο λόγια. Ο κύριος Λεφέβα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την έκθεση και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μαριά και τους υπολείπους για το περιεχόμενο. Αναγνωρίζουμε ότι σε καιρούς που αυξάνεται η δυσπιστία των πολιτών προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η Επιτροπή σας διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αναφέρεται άλλωστε και στην ε, έκθεση στο σχέδιο έκθεσης, διότι αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων. Προσωπικά έχω σταθεί σε τρία σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι το λεγόμενο τέρας του Λόχνες θα έλεγα, το θέμα της ερμηνείας του άρθρου 51 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι μια ιστορία χωρίς τέλος αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκανθεν εφάρμοζε την ομολογία του δικαστηρίου. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Επομένως, ε, δεν υπάρχει ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, ε, αλλά ε, το θέμα είναι σε επίπεδο κρατών μελών ή σε άλλο επίπεδο για το κατά πόσον θα αλλάξει αυτό το άρθρο και κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να αλλάξει. Ένα δεύτερο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχει σχέση με το Brexit και τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση και θα πρέπει να ε, το λάβουμε υπόψη, να δούμε όλα τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών ή και Βρετανών πολιτών που θα μείνουν στην Ευρώπη μετά το Brexit και ασχολούμαστε πισταμένα με το θέμα αυτό, όπως γνωρίζετε. Το τρίτο είναι η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών, ε, όπως ε, είδατε υπάρχουν προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βελτιωθεί αυτό το σημαντικό εργαλείο και να ε, προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε και την πρόσβαση, αλλά επίσης να υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα για προτάσεις δηλαδή οι οποίες ε, θα γίνουν λόγω ε, μελλοντικών πρωτοβουλειών πολιτών. Τέλος, ο κύριος Μαριάς αναφέρει στην έκθεση ότι εκτιμά το έργο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Ε, το ίδιο κάνουμε και εμείς και πιστεύουμε ότι η παρούσα Διαμεσολαβήτρια, η κυρία Οράιλη, κάνει εξαιρετική δουλειά και ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα, θα το φανταστείτε άλλωστε, ότι πέρσι ε, πρότεινε και το βραβείο αυτό της χρηστής διοίκησης, διότι αυτή δεν είναι μια διαδικασία στην οποία απλώς κατηγορούμε ε, αλλήλους, αλλά πρέπει να συγχαίρουμε και από καιρού καιρούν και ε, ήταν πολύ ευπρόσδεκτο αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν ε, για τη δουλειά σας. Θα παρακολουθήσουμε και την ψηφοφορία και το αποτέλεσμα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την επικοδομητική συνεισφορά σας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω και να ενισχύσουμε τη διοργανική συνεργασία και νομίζω ότι πλέον βρισκόμαστε πιο κοντά ε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι το εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτά. Ευχαριστώ. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 18 Οκτωβρίου, την επόμενη Τετάρτη στις 3 η ώρα. Και τώρα ε, θα αποχωρήσω και ο κύριος Σάκη θα συζητήσει το επόμενο θέμα. Να δώσω όμως αμέσως το λόγο σε εσά κύριε Μαριάν, ε, να ζητήσω συγγνώμη όμως διότι πρέπει να φύγω σε μια άλλη συνεδρίαση. Ιδιαίτερα σύντομα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους, οι οποίες βεβαίως θα ληφθούν υπόψη. Ε, να επισημάνω ότι στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων αναφέρομαι σε αυτό που έγινε το 2016 διότι η έκθεση δράσης της Επιτροπής αφορά το 2016. Άρα λοιπόν το σημείο 16 στο οποίο αναφέρομαι είναι εντός του πλαισίου. Τώρα το αν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις ή συνάλφοι που διαφωνούν αυτό είναι ένα άλλο θέμα και προφανώς ε, μπορούν να διατηρήσουν την άποψή τους. Ε, επίσης, ε, να πω στην κυρία Βαλίνα, προφανώς και γνωρίζω ότι το Σεπτέμβριο του 2016 η ΓΚΟΕ ψήφισε την πρότασή μου και αυτό το έχω πει και δημόσια, αλλά δυστυχώς σήμερα πριν λίγο στους συντονιστές η ΓΚΟΕ ψήφισε μαζί με τις άλλες δυνάμεις ενάντια στην πρότασή μου για διενεργία δημόσιας ακρόασης φέτος για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Εγώ εκτιμώ τη, τη θέση του κ. Τζάκη, ο οποίος λαμβάνει υπόψη το εξής ότι και στη χώρα σας υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά από το 1947 και υπάρχει και μία ε, αναφορά η οποία λέει τι θα γίνει με τις περιουσίες το 1947, ο περίφημος κανόνας Μπένες. Άρα λοιπόν βλέπω ότι τα θέματα του παρελθόντος όταν φτάνουν μέχρι σήμερα προφανώς δεν έχουν κλείσει και κάποια στιγμή θα κλείσουν. Εγώ είμαι αισιόδοξο σε πολύ πιο σύντομο διάστημα. Ελπίζω σε αυτή τη θητεία ή στην επόμενη να έχουμε μια θετική λύση επί του θέματος αυτού που είναι σοβαρό όπως είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις. Να πω όμως το εξή. Από τη συζήτηση προκύπτει και ήθελα να κάνω μια πρόταση προς τους συναδέλφους και στην Πρόεδρο η οποία θα τη λάβει υπόψη. Ε, πράγματι έχουμε λίγους αναφέροντες οι οποίοι έρχονται εδώ για να υποστηρίξουν την αναφορά τους. 61 πρόσωπα άτομα είναι λίγα. Και έρχονται λίγοι διότι υπάρχει το θέμα το οικονομικό. Δεν έχουν τα χρήματα να έρθουν στην Επιτροπή, υπάρχουν έξοδα, είναι μια εποχή δύσκολη με φτώχεια και ανεργία. Προτείνω μήπως θα μπορούσαμε να γίνεται συζήτηση με τηλεδιάσκεψη Δηλαδή έχουμε όλα τα μέσα εδώ στην Επιτροπή μας και θα μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι, οι αναφέροντες, στα γραφεία της Επιτροπής είτε της Κομισιόν, είτε στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη-μέλη, είτε σε άλλο χώρο, να συμμετέχουν στη συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης. Αυτό θα είναι πολύ πιο σημαντικό και με αυτόν τον τρόπο βεβαίως ε, θα έχουμε την άμεση παρουσία τους. Ήδη σημαντικές αποφάσεις με τηλεδιάσκεψη λαμβάνονται υπόψη στο Eurogroup και καταλαβαίνετε ότι μπορούν να υπάρχει συμμετοχή και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Εγώ μένω στο σημείο αυτό. Δεύτερον, σε σχέση με την Κομισιόν να πω ότι η Επιτροπή μας είναι αυτή η οποία ανοίγει τα θέματα και έτσι λαμβάνει γνώση και η Κομισιόν για να ασκήσει την διαδικασία παραπομπής ενός κράτους μέλους για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Θα λάβω υπόψη τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και περιμένω τις τροπολογίες για να δούμε ε, σε ποια θέματα θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Από ό,τι φαίνεται στα περισσότερα ζητήματα λίγο ως πολύ έχουμε συμφωνήσει. Υπάρχει αυτό το γνωστό θέμα που διχάζει την Επιτροπή. Θα εμείνω στην άποψή μου για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Προφανώς και εσείς και από εκεί και πέρα με δημοκρατικό τρόπο όπως είπατε θα βγει μια απάντηση αλλά ιστορικά θα μείνει ανοιχτό το θέμα αυτό όσο δεν το λύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσοι είναι αρμόδιοι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαριά. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό και μας λείπει άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η δική μου προφορική έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στη Λάρνακα της Κύπρου. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, ε, τη γραμματεία, τους εμπειρογνώμονές μας καθώς ε, και ε, τους ανθρώπους ε, στην Κύπρο. Ήταν πολύ καλή η διοργάνωση της επίσκεψης και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέρφους. Είχαμε πολύ καλή ομάδα. Δύο προβλήματα είχαμε. Το πρώτο είναι η ακτή και το λιμάνι της Λάρνακας, ε, ε, διότι κοντά στην ε, ακτή μήκους 1,5 χιλιόμετρου υπάρχει λιμάνι που χρησιμοποιείται και για βιομηχανικούς σκοπούς και οι πολίτες υπέβαλαν αναφορά διότι φοβούνται ότι εκεί ε, μεταφορτώνονται και ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Εξετάσαμε λοιπόν πολύ σοβαρά την κατάσταση στη Λάρνακα. Την δεύτερη μέρα ήμασταν στην Λευκοσία, όπου διαπιστώσαμε πόσο διαφορετικές απόψεις έχουν ε, μεταξύ τους τα διάφορα Υπουργεία για το ίδιο θέμα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πολύ καλός συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων. το Υπουργείο Οικονομικών μας ενημέρωσε ότι έχει προγραμματιστεί η κατασκευή νέου λιμένα όπου θα μεταμορφώνονται οι επικίνδυνες ουσίες, ενώ το λιμάνι το υπάρχον θα χρησιμοποιείται μόνο για τουριστικούς σκοπούς. Ε, αυτό φαίνεται να είναι επαρκής λύση και για την πόλη και για τους πολίτες. Ε, το άλλο πρόβλημα ήταν η βιομηχανική περιοχή κοντά στη Λάρνακα, όπου οι πολίτες ε, φοβούνται ότι χρησιμοποιούνται επικίνδυνες χημικές ουσίες. Εμείς δεν διαπιστώσαμε κάτι τέτοιο Πρέπει όμως ε, φυσικά να λάβουμε υπόψη μας σε τις ανησυχίες των πολιτών. Θα υποβάλουμε λοιπόν ε, τις συστάσεις για αυστηρή τήρηση των αδειών που παρέχει το Υπουργείο ε, και μας έχει διαβεβαιώσει και το Υπουργείο ότι δεν θα δώσει καμία άδεια για επικίνδυνες χημικές ουσίες. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα της ε, επίσκεψης. Ε, ο δήμαρχος της Λάνακας μας είπε ότι πρώτη φορά συναντήθηκε με εκπροσωπούς του λιμανιού όταν ε, ήμασταν εμείς εκεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μας και θα υποβάλουμε και γραπτό την έκθεση και το αργότερο τον Δεκέμβριο θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση. Ε, ρωτώ εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Από ό,τι βλέπω όχι. Σας ευχαριστώ. Α, και όμως, παρακαλώ. Ε, Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τα συγχαρητήριά σας. Πήγε πολύ καλά αυτή η επίσκεψη, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την οργάνωση, την Αταλία και τους άλλους. Ήταν εξαιρετική η επίσκεψη αυτή. Νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες αποστολές τις οποίες έχουμε κάνει. Θα συμφωνήσω με τα σχόλια τα οποία είπατε σε σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα γίνει με θέματα όπως ε, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα αρμόδια υπουργεία και μια δυσκολία, για να μην πω πλήρης, έλλειψη δυνατότητας επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν το πρωινό τμήμα της συνεδρίασης. Καλή όρεξη σας εύχομαι και θα συνεχίσουμε στις 2.30. Σας ευχαριστώ.